Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με την ημερησία μας διάταξη και τις ψηφοφορίες μας. Μετά από το πρωινό μαραθώνιο και ένα μικρό μαραθώνιο σήμερα το πρωί, πολύ σημαντικά θέματα στην ημερησία διάταξη. Σημείο 12 πρότυπα ποιότητα και ασφάλεια των ανθρωπίνων οργάνων που βρίσκονται για μεταμόσχευση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα. Εισηγητή ο Μύροσλαβ Μικολάσικ. Ο εισηγητή ήθελε σύντομα να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Sie haben das Wort. Ja. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να τονίσω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις και τη γραμματεία όταν προετοιμάσαμε το κείμενο και φτάσαμε σε μια πολύ καλή συνεργασία και συμβιβασμούς. Και από πλευράς εισηγητή θα ήθελα να πω ότι έλαβα υπόψη έναν ικανό αριθμό των ε, τροπολογιών σας, συνάδελφοι, όχι μόνο των σκιωδών, αλλά και άλλων που υπέβαλαν τροπολογίες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι έχουμε ένα κείμενο υψηλής ποιότητας σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Επίσης, είχαμε ένα θετικό ε, μήνυμα από την νομική υπηρεσία, το έχετε στο φάκελό σας και μπορώ να διαπιστώσω ότι το άρθρο 168 της οδηγίας μας δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουμε και ε, Επίσης μπορούμε να προωθήσουμε θέματα δωρεάς για μεταμόσχευση και ε, από πλευράς δωρητή, διευκολύνοντας την πλευρά του δωρητή. Θα ήθελα να μην υπάρξει παρεξήγηση σε σχέση με την ενοποιημένη, παγιοποιημένη τροπολογία 4, όπου έχω όλα τα στοιχεία του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί έγινε ε, μία δημόσια συζήτηση για την ενζωή δωρεά οργάνων. Νομίζω ότι η... χωρίς αυτήν την τροπολογία δεν θα είχε καν αρχίσει η συζήτηση σε αυτές τις χώρες, αλλά θα ψηφίσουμε και θα ήθελα να με υποστηρίξετε, διότι το Κοινοβούλιο έχει θετική στάση, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρο το Κοινοβούλιο και έχουμε και μία όθηση από τα κράτη-μέλη που θέλουν να εγκριθεί αυτή η οδηγία το ταχύτερο δυνατόν. Άρα, ε, όχι μόνο η σημερινή ψηφοφορία, αλλά και η τελική ψηφοφορία το Μάιο στο Στρασβούργο θα ε, θα μας ε, οδηγήσει στο να διαθέτουμε αυτή την οδηγία σύντομα για τους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Νικολάουσικ. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 59. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung beendet. Πέρασε ψηφοφορία. Α, 27 υπέρ, 18 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Μετά. Τροπολογία στην επόμενη σελίδα 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64-65 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 72 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέξουμε. Check, check. So, beendet. Ja, Απερίφθη πράγματι. 74 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και εδώ. 74. und beendet. 28 zu 24. 28 προς 24, εγκρίνεται λοιπόν. Ε, 75, υπέρ. Κατά. Άποχες, παρέπτεται. 76, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 Τώρα τι κάνουμε. 77 ähm, 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 και 82 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε καλώς ελέγχουμε την 6 Πέρασε φορέ. 34 υπέρ, 19 κατά. Ναι, ναι, ξεκάθαρο ήταν. Ναι. Επόμενη σελίδα. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε. 87 ελέγχουμε. Α, έχει ψηφοφορία. Abstimmung geschlossen. Sure. Πέρα Το κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο. Απορρίπτεται. 26 προς 26. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 και 94 τώρα. μας Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 95. Υπέρ. κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά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 Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε. 108 ελέγχουμε. Άχι ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες Εγκρίνεται 28 προς 23. 110. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ αν Α, ναι, και 115 που είναι συμβατή μπορούμε να την ψηφίσουμε. Λοιπόν, 115, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. απεχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. απεχές απορρίπτεται. 118 με μία προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απερίφθη, αλλά για να το ελέγξουμε. Την 119 ελέγχουμε. Ε, ε. Πράγματι απερίφθη. Ναι, ναι, 20 προς 31. 120, υπέρ. Κατά άτοχες εγκρίνεται. 121, υπέρ. Κατά άτοχες εγκρίνεται. Γιούρι 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. 139 να ελέγξουμε. Α, όχι, την 138. 138 να ελέγξουμε. Abstimmung beendet. Πολύ σαφέ. 50 προ 6. Ξεκάθαρο. 139 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 140 και 141 Ταυτόσιμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145-146 υπέρ. Κατά αποχές για να ελέγξουμε 145 146 ελέγχουμε πέρα ψηφοφορίας ψηφοφορίες ναι πραγματικά δύσκολο 29 προς 28 εγκρίνεται όμως 23, ζούρι 5 και ζούρι 4. Όχι. 23 και ζούρι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ζούρι 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 και 148. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 24 καταπίπτει. 150 συνεχίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι είναι σαφές. Για να ελέγξουμε. Για την 150 ελέγχουμε. und beendet. Πέρας. Ναι, 28 προς 26. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Τη 25 να τα ελέγξουμε. Πέρασε. 32 υπέρ 22 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επόμενη σφίδα. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 και ζούρι 8 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 και ζούρι 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ζούρι 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157-158 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Μάλλον ενοποιημένη. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Έχει την ψηφορία για την ενοποιημένη τροπολογία περιθμών 4. Πέρας ψηφοφορία. Α, έγινε δεκτή. 31 προς 24. 162. Υπέρ. Σελίδα 17. 162. Υπέρ. Κατά. Για να δούμε. Για να το ελέγξουμε. 162. Σειρά 17. Also, Abstimmung ist geschlossen. Doch klar, 34 dafür. 34 kata, engrinete. κατά εγκρίνεται. Dann ganz unten auf Seite 17 168. 168 πάντα σελίδα 17 υπέρ. Dagegen. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 34, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Ξανά, 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απερίφθη, αλλά για να το ελέγξουμε. 179. Abstimmung geschlossen. Πέρασε Ναι, ξεκάθαρα περίφθη. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 και 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 184 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 και 191 ε, ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 192 και 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Την 197 ελέγχουμε. Ένα από το ΕΚ. Περισσεύει. Ακόμα. Εντάξει. 29 υπέρ 27 κατά. Είναι κρίθη λοιπόν. 49 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κυρία Άση, προφορική τροπολογία για την 54. Έχω μία προφορική, αγαπητή συναδελφή έτσι ώστε αυτό το θέμα να συμβαδίζει με την πρώτη έκθεση του Γιολάινεν, την οποία ψηφίσαμε σήμερα το πρωί. Στην πρώτη παράγραφο το κείμενο θα λέει επεκτείνεται κατά ένα μήνα, αντί για, για δύο μήνες αντί για ένα μήνα, όπως αποφασίσαμε σήμερα το πρωί. Ωραία, δεν διαφωνεί κανένα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν με αυτή την προφορική τροπολογία για το 54. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Βέβαια, να συμφωνείτε με τον πρόεδρο πάντα είναι πολύ καλό. 55 dafür. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200 και 201 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 56, 202 και ζούρι 11. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο τελικές ψηφοφορίες. Καταρχήν για το σχέδιο έκθεσης ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ένας από το ΕΛΚ είναι περισσότερος από ό,τι πρέπει. Ο άλλος είναι Εντάξει τώρα. Λοιπόν, 56 προς 0 προς 1. Συγχαρητήρια. Και τώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα. 53 προς 0 προς 1. Συγχαρητήρια τον συνάδελφο Μικολάσικ. Την επόμενη εβδομάδα στη μεγάλη διάσκεψη στη Μαδρίτη, τη Διεθνή Διάσκεψη για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, θα μιλήσετε στην έναρξη και θα είναι παρούσα και μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. I, I just to... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι μας καθοδηγήσατε σε αυτή την ψηφοφορία και σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα στη διάσκεψη της Μαδρίτης την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα υποφεληθούν στην Ευρώπη από αυτά που αποφασίσαμε και ψηφίσαμε. Και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Που και αυτό έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Την έκθεση του Ανδρές Περέλο Ροντρίγκες. Και περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Για την 10. Check Πέρας. 24 προς 33. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 3. Υπέρ. Αν δεν θα ψηφιστεί αυτή βλέπω. Περνάμε στη 13 λοιπόν. Τρο... Ε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 1 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Γιούρι 2 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Για την ε, Γιούρι 5, παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. And the Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Α, συγγνώμη, ενοποιημένη, κωδικοποιημένη 2 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό αν θέλετε. Έναρξη ψηφοφορίας. Abstimmung geschlossen. Πέρας. 29 26. 29 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. Και περνάμε στην 24 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 9, υπέρ. Κατά. Αποχές Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Για την Γιούρι 9. Abstimmung beendet. Πέρας. Καλά το είδατε. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη υπαρθμό 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 31 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 7. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αποσύρεται η 1, Γιούρι Α τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι Β, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η πέντε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορίας, παρακαλώ. Είναι πιστικό το αποτέλεσμα. 58 ψήφοι υπέρ και καμία ψήφος κατά. Μία αποχή. Να συγχαρούμε τον συνάδελφο για την έκθεση και την ε, δουλειά που έκανε.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 Punkt Nummer 14, gemeinsam durch στο 14 το κοινό πρόγραμμα Έρευνα και ανάπτυξη στη Βαλτική θάλασσα. Το πρόγραμμα Bonus, Όπω ονομάζεται, η Άννα Ροσμπαχ είναι η συγγήτρια και θα περάσουμε στην ψηφοφορία τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 21 υπέρ. 21 και 22. Συμβατές και ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είδα να σηκώνουν τα χέρια οι φιλελεύθεροι. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 21 και 22. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung geschlossen. Das war... Peras. Καλά κάναμε και το ελέγξαμε. 27 η ψήφη υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. Και περνάμε στις 23 και 25 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά Να το ελέγξουμε και αυτό αν θέλετε για την 23 και την 25 ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Και αυτή καλά κάναμε και την ελέγξαμε. 25 ψήφοι υπέρ, 24 κατά. 26 στη σελίδα 2, είπε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 και 33 είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 και η 40. Οι 38 και 40 καταπίπτουν. Η 41 τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία τώρα για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 54 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Να συγχαρούμε την εισηγήτρια για την έκθεση της αυτή για τη Βαλτική θάλασσα. Συνάδελφοι, είσαστε τρομεροί. Δεν χρειάζεται να πάτε καν στο γυμναστήριο με τόσε φορέ που έχετε σηκώσει το χέρι σα. Αλλά συνεχίζουμε ακάθεκτη στην επόμενη ψηφοφορία. Για τη λευκή βίβλο. Α, όχι, μισό λεπτό. Genau. Wir haben zuerst noch die Abstimmung über Punkt 15. Ψηφοφορία για το σημείο 15 για την κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η Τατσιάνα Οκτάβια Σάρμπου είναι η εισηγήτρια. Και περνάμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 αποσύρθηκε. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται η πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή της κυρίας Σόρμπου ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ Abstimmung geschlossen. Πέρας 51 ψήφοι υπέρ, 1 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Έχει προλιανθεί το έδαφος για μια ενεργειακά πολιτική οικονομία με την έκθεση αυτή. Και περνάμε στο σημείο που έπρεπε να έχουμε φτάσει στις 3 η ώρα στο σημείο υπαριθμών 16, λευκή βίβλος, η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης. Ο Βιτόριο Πρόντι είναι ο εισηγητής. Και έχουμε συμβαστικές τροπολογίες, ε, τις έχετε μπροστά σας. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Συμβαστική υπαριθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η υπαριθμόν 20 με μια προφορική τροπολογία από τον Μπάς Ικχάουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να προσθέσω την... Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και για τη δασοκομική πολιτική έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ΚΑΠ, η πολιτική αλίας, η δασοκομική, καθώς και μία μελέτη αντικτύπου ως προς τα περιβαλλοντικά. Δηλαδή, στην ουσία προσθέτουμε τη δασοκομική. Αποδεκτή η προφορική τροπολογία, να την ψηφίσουμε την 20 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε, λέει ο Πρόεδρος, για την 22. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung beendet. Πέρας. 27 προς 25 εγκρίνεται. Και περνάμε στην επόμενη σελίδα τώρα, στην 24, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται 25, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 30 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Το δεύτερο τμήμα της 30. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Abstimmung beendet. Πέρας. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 31 προς 21 εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 12 Α, 35, ε, συγγνώμη, 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέγγι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε για την 45. Ja, das war... Ναι, δίκιο είχα και το έλεγξα. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. Έχετε το λόγο, ναι. Δεν έχω την κάρτα μου, αλλά ψήφισα. Äh, äh, <laughs> ναι, κρίμα, αλλά χρειάζεστε την κάρτα σας για να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Έτσι έχουν ε, οι κανόνες μας. Τι να κάνουμε, λυπάμαι. Και προχωράμε. Συνεχίζουμε με την 46. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Πολύ λυπάμαι αγαπητέ συνάδελφε. Τι να κάνουμε, ονομαστική κλίση σημαίνει ονομαστική κλίση. Και περνάμε στη 48, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 49, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 52 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 60 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η 64 και η 65 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 64 και την 65. Έναρξη ψηφοφορίας.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 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 68 η 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία, για την 68. Abstimmung geschlossen. Πέρα Σαφή η πλειοψηφία υπέρ. Και συνεχίζουμε στην 74. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Υπέρ. Για την 74. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε για την 92 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας. Abstimmung geschlossen. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται 92. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαφές το αποτέλεσμα. Είναι σαφές, ε, Κρίστελ. 98 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επόμενη σελίδα 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέζι 17 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δεκαπέντε, Σίμπερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές κρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 128 ελέγχουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Να ελέγξουμε την 129. Abstimmung ένα Ενεκρίθη. Πολύ ωραία. Δεν σηκώνουν όλοι τα χέρια του πια γι' αυτό. 130 είμαστε τώρα. 130. Θεόδωρο Κυλακάκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 split 113 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 134. Abstimmung beendet. Ja. 26 dafür, 28 dagegen. Απορρίπτεται 26 προς 28. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18. Dafür. Ρεζί 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρεζί 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ρεζί 14 ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung beendet. Πέρασε πληροφορίε. πληροφορίες. Για ναι, ξεκάθαρα, 31 προς 23. Εγκρίνεται. Σουρι 2, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται. 143, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 144, υπέρ. Κατά. Απεχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Ρέτζι 15. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίες. Ναι, 36 προς 16 ξεκάθαρα υπέρ. Ρέζο 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 153 ε, να ελέγξουμε 152 να ελέγξουμε πέρας πληροφορίας καλά το είδα 26 προς 27 απερίφθη 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά Να ελέγξουμε. Την 155 ελέγχουμε. Πέρασε πληροφορίες. Ναι, ναι, πράγματι. Απορρίπτεται 27 προς 27. 156 υπέρ. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ζούρι 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε 161 να ελέγξουμε 30 υπέρ και 23 κατά. Εκατόν υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω, δεν σηκώνει το χέρι Λοιπόν, 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέζι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέζι 19 καταπίπτει. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτό Πολύ ωραία. Γιατί φτάνουμε σε τελική σκέψη, στη σελίδα 16. Πολύ ωραία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά αν θέλετε να το ελέγξουμε. 7. Πέρας ψηφοφορίας. Είναι κρίθη. 27 προς 20. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά.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 Ζούρι B. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται και ζούρι C. Γάμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Ζούρι ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Η ηλεκτρονικά την ε, νομοδότηση του Βιτόριο Πόντι. Άχι ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 49 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια τον εισηγητή. προσωμολογία είναι το δεύτερη ο δεύτερο πυλώνα για την προστασία του περιβάλλοντο. Εργαστήκαμε θαυμάσια συνάδελφοι. Τελώ την ψηφορία, αλλά συνεχίσει η συνεδρίαση. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Als da wäre Σημείο 17. ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για το οποία απαιτείται η ιατρική συνταγή. Κρίστοφερ Φιέλνερ είναι ο εισηγητής. Mr. Chairman, if it's okay, I'll wait a couple of minutes until... Θα περιμένω δύο λεπτά, έτσι ώστε να φύγουν όσοι είναι να φύγουν. That's better. Come here. Bien. Alors, pour les courageux qui restent... Για τους θαραλέους που παρέμειναν, θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ε, une information sur... Με μερικές ε, πληροφορίες για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, φάρμακα για τα οποία απαιτείται η ιατρική συνταγή. Δία, 2001 του 83, ο κύριος Φέλνερ μπορεί να λάβει το λόγο, αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά να αρχίσω την παρουσίαση αυτού του σχεδίου έκθεσης. Καταρχήν, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υφίσταται πρόβλημα. Να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε απαράδεκτες διαφορές στην πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ανισότητα μπορεί να δημιουργήσει και ανισότητα στο, στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας και θα ήθελα να πω σε αυτούς που δεν διαβάζουν αγγλικά ότι οι περισσότερες πληροφορίες ίσως δεν υπάρχουν στη μητρική τους. Επίσης υπάρχουν πολλές μη ελεγχόμενες πληροφορίες ιδιαίτερα στο ίντερνετ και είναι δική μας ευθύνη να είμαστε σίγουροι ότι είναι ελεγχόμενες αυτές οι πληροφορίες. Τέλος θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε τον αλφαβητισμό των ε, ασθενών σε θέματα υγείας. Γιατί χωρίς πληροφορίες ε, δεν μπορούμε να έχουμε την αντιμετώπιση των θεμάτων των πραγματικών ασθενών. Δεν έχουμε πλήρη απάντηση από το Κοινοβούλιο και όχι σε όλα τα μέρη. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος του παζλ, ένα πολύ σημαντικό η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να αλλάξει. Έχετε 40 σελίδες αλλαγών που πρότεινα και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε πέντε, στις πέντε σημαντικότερες. Καταρχήν, νομίζω ότι η πρόταση που λάβαμε από την Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη την οπτική ε, γωνία των ασθενών. Άλλαξα λοιπόν την οπτική γωνία, όχι δηλαδή της βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά των ασθενών. Δεν με ενδιαφέρει η θέση της φαρμακοβιομηχανίας. Με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των ασθενών, το δικαίωμα στη γνώση. Άρα προσπάθησα να αλλάξω ε, ορισμένες θεωρήσεις, ε, να μιλάμε για υποχρέωση παροχής ε, πληροφοριών και όχι διάδοση πληροφοριών. Και επίσης να δίνουμε πληροφορίες ζωτικής σημασίας. Αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στις δεσμίδες εγγράφων. Είναι ελεγχόμενες αυτές οι πληροφορίες όμως. Αυτό αφορά και τους διαφόρους ιατρικούς συλλόγους. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση πριν από την αδειοδότηση να ελέγχεται αυτή η πληροφόρηση. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα που θέλει διαφήμιση για συνταγογραφούμενα φάρμακα, διότι στις ΗΠΑ η κατάσταση δεν είναι κανόνας και δεν θέλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό προσπάθησα να ενισχύσω την απαγόρευση, απαγόρευση διαφήμισης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μιλάμε για ε, πληροφόρηση push and pull και το σκέλος push να μην υπάρχει. Μόνο όταν ζητούν πληροφορίες οι ασθενείς θα πρέπει να τους δοθεί πληροφόρηση. Αν δεν ζητηθεί δεν πρέπει να δοθεί. Επίσης, δεν λαμβάνω υπόψη τις πληροφορίες μέσα από περιοδικά υγείας. Άρα τηλεόραση, ΜΜΕ, τύπος, όλα αυτά δεν θα είναι ένα κανάλι πληροφόρησης. Μόνο όταν ζητείτε η πληροφόρηση θα ε, δίδεται, θα χορηγείται. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η αρχική πρόταση δεν αφορά τη συμμετοχή των ασθενών. Γι' αυτό θα ήθελα να συμμετέχουν και οι ασθενείς και οι φορείς Υγεία στην εφαρμογή της οδηγίας, έτσι ώστε να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Για να ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα για την προώθηση της απαγόρευσης. Δεν θα πρέπει να διολυσθένει ε, κάποιο είδος πληροφόρησης, δεν πρέπει να προωθήσουμε κανένα είδος διαφήμισης. Γι' αυτό οι φορείς υγείας και οι ασθενείς θα πρέπει να εποπτεύουν την τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών γιατί είναι, αυτοί είναι οι άμεσα ευεργετούμενοι από την πρόταση, γι' αυτό πρέπει να συμμετέχουν και στην κατάρτισή της. Ε, εάν τώρα υπάρχει κάτι το οποίο δεν υπησέρχεται στην πληροφόρηση και θα ήθελα να αναφέρω, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία διάρθρωση εποπτείας για κυρώσεις όπου να συμμετέχουν και ασθενείς και χωρίς υγείας, έτσι ώστε να βλέπουμε αν υπάρχουν παράπονα, να διοχετεύονται και έτσι ώστε όποιος δεν συνδράμει σωστά να τιμωρείται. Θα επανέλθω σε αυτό αν βρω την καλή διάρθρωση, αλλά είναι κάτι που δεν υπάρχει στην πρόταση. Με απασχόλησε όμως, δηλαδή να υπάρχει μία διάρθρωση παραπόνων που υπάρχει στη Γερμανία στον τομέα της διαφήμισης. Εάν δει κάποιος κάτι το οποίο είναι εσφαλμένο, μπορεί να προβάλλει ε, συγκεκριμένα παράπονα, κάνει προσφυγή κατά της διαφήμισης. Το τέταρτο σημείο είναι ότι προσπάθησα να διασαφηνίσω την εμβέλεια της ε, οδηγίας, διότι έχουμε και προσφυγές σε εθνικά δικαστήρια Δηλαδή είδαμε ότι δημοσιογράφοι ε, επέκριναν αυτή την διάρθρωση και θα πρέπει να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Οι δημοσιογράφοι, οι ασθενείς, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκφράζουν, δηλαδή να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους για τα φάσμακα. Φάρμακα, τα φαρμακευτικά σκευάσματα γι' αυτό, κατέστησα σαφές ότι αυτός ο κανονισμός δεν αφορά αυτούς τους φορείς. εκτός αν δρούν εξ ονόματος της φαρμακοβιομηχανίας. Αν δρούν αυτόνομα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Τέλος, τόνισα ότι το πιο, ο πιο σημαντικός διάβλος είναι ο ιατρός που συνταγογραφεί. Οποιοδήποτε άλλος διάβλος θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται συμπληρωματικά στοιχεία, διότι ε, ένας ασθενής βρίσκεται ενώπιον του γιατρού για 5 με 7 λεπτά πριν του συνταγογραφηθεί ένα φάρμακο και πολλές φορές ορισμένα ε, δελτία χάνονται, ενημερωτικά δελτία. γιατί πολλές φορές δεν τα λαμβάνουν υπόψη οι ασθενείς ή δεν μπορούν να δώσουν συνέχεια. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πέντε σημεία στα οποία εστίασα την προσοχή μου και καταλαβαίνω ότι μερικοί συνάδελφοι ρώτησαν κατά πόσο δεν θα έπρεπε να αναβάλουμε το όλο ε, εγχείρημα. Στην ακρόαση του κυρίου Ντάλι ελέγχθη ότι ίσως αναθεωρηθεί η πρόταση. Διαφωνώ όμως, γιατί είναι δική μας δουλειά να προβάλλουμε την αναθεώρηση και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να αναθεωρήσει την πρόταση, δεν θέλω να βασιστεί σε αυτά που είπε το Συμβούλιο και μόνο. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα και προέβαλε ορισμένες δηλώσεις. Θα πρέπει όμως να ακουστεί και η δική μας φωνή. Εάν λοιπόν υπάρξουν ε, περαιτέρω προτάσεις από την Επιτροπή, θα πρέπει να προβάλλουμε τη δική μας άποψη. Αυτό θα ήθελα να το καταστήσω σαφές. Θα ήθελα να ε, ζητήσω, μάλλον να ευχαριστήσω και τους βοηθούς που με συνέδραμαν και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, οργανώσεις και ενώσεις ασθενών για το input. Εμπνεύστηκα από τις συναντήσεις μας. Τώρα προσμένω τη συνεργασία μαζί σας. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα. Όλα είναι στο σφυρί. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας εκτιμήσεις. Euh, σας ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Ο πρόεδρος, ο κύριος ε, Περέλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι ο κύριος ε, Περνό ε, ήταν σκιώδης, αλλά έπρεπε να φύγει. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική μας θέση. Σε αυτή την Επιτροπή γίνονται θέμα συζητούνται θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης και καταπολέμησης της ε, απάτης των φαρμακοσκευασμάτων και μας ενδιαφέρουν και οι μελλοντικές προσδοκίες σε αυτό το τομέα. Αλλά δυστυχώς ξεχνάμε πολλά στοιχεία και πολλές φορές δεν συνδράμουμε τους ασθενείς. Η κοινωνία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να υπερασπιστούμε, να προστατεύσουμε τους ασθενείς. Είμαστε σκεπτικοί έναντι της φιλελευθεροποίησης, της τάσης φιλελευθεροποίησης που διαγράφεται ε, στο έγγραφο βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η ζωή των πολιτών και θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Άρα, όταν μιλάμε για αλλαγή κανονιστικού πλαισίου για να έχουν άμεση πρόσβαση οι ασθενείς στα νέα σκευάσματα, θα ήθελα να πω ότι δεν δεχόμαστε το σημείο εκκίνησης. Το σημείο εκκίνησης. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό αίτημα ούτε από τους ασθενείς, ούτε από τις αρχές, ούτε από τους ιατρικούς φορείς. Κανείς δεν ζήτησε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η πείρα μας μας δείχνει το εξής, ότι ο πολίτης έχει πρόσβαση σε σωρία πληροφοριών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να κρίνει μία φαρμακευτική καινοτομία, γιατί σε δίνει σε θέση. Ο τομέας υγείας παρέχει σωρία πληροφοριών αλλά οι πληροφορίες προς τον ασθενή είναι ένα θέμα που αφορά τον επαγγελματικό κλάδο, δηλαδή τον ε, τομέα υγείας και τα εθνικά συστήματα υγείας. Γι' αυτό θα ήταν λάθος να υπερβάλλουμε το κόστος πληροφόρησης χωρίς να υπάρξει κανένα πλεονέκτημα για την προστασία της υγείας. Έχουμε μπροστά μας μία πολύ σημαντική εργασία στο πακέτο φαρμακευτικών σκευασμάτων. Άρα θα πρέπει να ρυθμίσουμε το πλαίσιο μόνο εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το πακέτο της Κομισιόν δεν ενέχει τα κατάλληλα στοιχεία για να καταρτήσουμε μια σωστή οδηγία. Και θα ήθελα να πω απλά ότι το κείμενο αυτό μας δείχνει ότι στοιχίζει περισσότερο να αλλάξουμε αυτή την οδηγία από το να συγκροτήσουμε, να συγγράψουμε μία καινούρια. Δεν ε, κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν να αναθεωρηθεί, διότι το ενεχόμενο κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό και δεν χρησιμεύει κατ' ουσίαν. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φιέλνερ, γιατί συζητάμε εδώ και καιρό το θέμα αυτό. Και είπε ακριβώς αυτά που απαντούν στον συνάδελφο Ντεγκράτο που είπε ότι θα πρέπει να αναπέμψουμε το θέμα αυτό. Αλλά, συνάδελφε, αυτή είναι η δουλειά μας, να αλλάζουμε τις ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το έργο μας. Δεν μπορούμε να τα αναπέμπουμε όλα και ο κύριος Φιέλνερ ανέφερε τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε προκειμένου να καταστεί το κείμενο αποδεκτό και από την ομάδα σας. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλή η πρόταση για την ε, αναπομπή του θέματος. Το εκρηκτικό υλικό, αν θέλετε, το οποίο υπήρχε στην αρχή, επειδή υπήρχαν κάποιες ηθελημένες παρανοήσεις, έχουν αφαιρεθεί. Ναι, δίκιο έχετε μεν. Αυτά τα ευαίσθητα συστήματα, αυτές οι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι στα χέρια εκείνων που είναι αρμόδιοι. Αλλά αυτό κάνει ο Κρίστοφερ Φιέλνερ με την έκθεσή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει λοιπόν μια νέα διαμόρφωση ενός ενήλικου ε, ευσυνείδητου ε, και ε, ασθενούς, ο οποίος μπορεί να σχηματίσει από μόνος του μια ιδέα και ο οποίος θα έχει πραγματικά σωστές πληροφορίες στη διάθεσή του, γιατί αυτή θα είναι η συμβολή μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπάρχει μια, ένας έλεγχος εξάντε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές σε κάθε κρατος μέλος, οι οποίες, ε, έλεγχος ο οποίος θα δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στον ασθενή στις σωστές πληροφορίες. Άκουσα ότι κάποιοι συνάδελφοι, οι πράσινοι, θέλουν να αναβληθεί η ψηφοφορία. Να σας πω ότι συμφωνώ με τον Επιτροποντάλη, ο οποίος είπε ότι από πλευρά του Συμβουλίου έχω πλέον την τοποθέτηση του Συμβουλίου μπροστά μου, θέλω να μάθω και ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι και το, τη δυνατότητα έχουμε και την ευθύνη έχουμε να παρουσιάσουμε τη δική μας θέση από την ε, Επιτροπή Βιομηχανίας ως εισηγητής. Θα ήθελα να περιοριστώ σε περιορισμένα σημεία. Αυτό που δημιουργήσαμε για να δημιουργηθεί ένα σημείωμα και με τις τροπολογίες που προτείνει ο κ. Φιέλνερ έχουμε τη δυνατότητα καταρχάς να έχει μια κατανοητή μορφή αυτό το σημείωμα το οποίο επισυνάπτεται στο φάρμακο. Να υπάρχει τυποποιημένη μορφή, κατανοητή σε όλες τις γλώσσες και να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Αυτή είναι ε, η ουσία των όσων προτείνει ο κύριος Φιέλνερ και νομίζω ότι σε μια εποχή που ο κόσμος ταξιδεύει και δεν κουβαλάει μαζί του αυτά τα χαρτιά θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρχουν πιστοποιημένες πληροφορίες εξάντε. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Ναι. Τέθηκε και το ερώτημα του ποιοι σε δι θα χρησιμοποιηθούν. Έχουμε καταρχάς τις ε, διόδους, αν θέλετε, που αφορούν τη δημόσια υγεία, αλλά, συνάδελφε, δεν συμφωνώ με την ε, πρόταση αναπομπής. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει, να μην επιτρέπονται οι διαφημίσεις. Και αυτό, ε, γι' αυτό αγωνίζονται επειδή επί σειρά ετών πολλοί κόσμος δεν επιτρέπονται αυτές οι διαφημίσεις σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. όπου επιτρέπεται αυτό από το Σύνταγμα. Θεωρώ ότι τρέχουσα συζήτηση πραγματικά δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της εποχής μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είναι σημαντικό για τον κόσμο στην Ευρώπη. Η υγεία του. Θα πρέπει να το λάβουμε πιο στα σοβαρά και να δώσουμε πιο μεγάλη ευθύνη στον κόσμο και να μην ξεχνάμε ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει την πιστοποίηση αυτή για τα κεντρικά, αν θέλετε, επιστοποιημένα φάρμακα θα είναι η ΕΜΕΑ αυτή η υπηρεσία που εδρεύει στο Λονδίνο. Είναι ευρωπαϊκή υπηρεσία και η ΕΜΕΑ χρειάζεται πιο πολλά κονδύλια και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να τους επιβάλλουμε να, να κάνουν πιο πολλή δουλειά και να μην τους δίνουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα. Και πάλι να επαναλάβω ότι χαίρομαι που δεν αποσύρει την πρόταση αυτή ο Επίτροπος Ντάλι και ευχαριστώ και πάλι τον συνάδελφο Φιέρνερ, ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ υπομονετικά. Merci, Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Χάση για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω την διαδικασία μαζί σας, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε την νομοθετική διαδικασία που προβάλλεται στο Κοινοβούλιο, διότι ο Επίτροπος Ντάλι, όταν παρευρέθηκε σε αυτή την Επίτροπη, δεσμεύθηκε να επανεξετάσει αυτή την πρόταση, διότι και επειδή ακριβώς είναι παρόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδιατυπώσει αυτή την πρόταση ή όχι. Και μετά την απάντηση της Επιτροπής θα επανέλθω. Uh, είναι έτοιμη να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλει να απαντήσει η Επιτροπή, παρόλο που δεν είναι η τρέχουσα διαδικασία, μπορεί. Μόνο σε αυτό το ερώτημα, γιατί επί του συνόλου θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Ο Επίτροπος Ντάλι όντως ε, στην ακρόαση, στην Επιτροπή σας αυτή, είπε ότι θέλει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση τροποποίησης και ότι θέλει να τονιστεί η διάσταση του ασθενού σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή, αλλά να μην παρεξηγήσουμε να μην θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μία ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα υποβάλει, υποβάλει μάλλον μία τροποποιημένη πρόταση και επιθυμεί να διακοπεί η θεσμική διαδικασία. Αντιθέτως, ο Επιτροπός Ντάλι σκοπεύει στο σημείο αυτό να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής αυτής να μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι οι δηλώσεις του υπονοούν ενδεχόμενη διακοπή της θεσμικής διαδικασίας. Ευχαριστώ και ελπίζω αυτό με διευκρινίζει κάπως την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάση, αν θέλει να θέσει άλλο ερώτημα. This clarification. Uh, anyway, uh, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την διευκρίνηση. Ο Επίτροπος Ντάλι είπε ότι θα λάβει υπόψη την απτική γωνία των ασθενών καταρχήν και μετά θα γίνουν οι κατάλληλες, οι δέουσες συζητήσεις μαζί σας. Άρα το Κοινοβούλιο έχει τον κανόνα υπαριθμό, το άρθρο 53 του κανονισμού που λέει ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώσει την Επιτροπή ή εάν ε, η εμπλεκόμενη Επιτροπή μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιεί την πρότασή της, η ενδιαφερόμενη Επιτροπή θα αναβάλει την εξέταση μέχρι ότου λάβει μια νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη εργασία για μας, αν πρόκειται για ένα καθαρά νομοθετικό έργο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια νέα συλλογιστική στην Επιτροπή και το θέμα αυτό το, ε, το έχετε μπλοκάρει, έχει μπλοκαριστεί μάλλον στο Συμβούλιο. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε, να μιλήσουμε να προβάλλουμε τη γνώμη μας στην Επιτροπή. Υπάρχει βεβαίως και η μη νομοθετική διαδικασία, η οποία είναι πιο εύκολη. Αν όμως ε, πρόκειται για μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, τότε θα έχουμε πολλές διαπραγματεύσεις επί θεμάτων τα οποία εξαφανίζονται Άρα νομίζω ότι οι συντονιστές θα πρέπει να ασχοληθούν με το ζήτημα, δυνάμει του άρθρου 53, και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν εναλλακτικέ. για να γνωμοδοτήσουμε και ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πριν έχουμε την ε, ε, τελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να αντικατοπτρίζει και την άποψη του Επιτρόπου. Άρα, για να είμαι σαφής, η πρότασή μου είναι να μην αποφασίσουμε, να μην ορίσουμε προθεσμία υποβολής τροπολογιών σε αυτή τη φάση. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιχειρήσω να γεφυρώσω αυτά που είπαν οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές, ο κύριος Κοντζημαρκάκης αφενός και αφετέρου ο Άντρες Περίεβιο και η Σάτου Χάση από την άλλη. Και σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Κρίστο Φιέλνερ γιατί πολλά ε, από αυτά που χρειάζονται για να γεφυρωθεί ε, η διαφορά αυτή περιλαμβάνονται στην έκθεση του, στο σχέδιο έκθεσης. Νομίζω και να το τονίσουμε αυτό ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως την έχουμε μπροστά μας σήμερα, χωρίς τις τροπολογίες του Κρίστοφερ Φιέλνερ, δεν προκαλεί μόνο παρανόηση, αλλά είναι πραγματικά κακή, κακίστη και όσοι ασκούν κριτική στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο γιατί αυτή η πρόταση της Επιτροπής δεν θα πρέπει να εγκριθεί όσο έχει. Αλλά αφετέρου να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για μας, για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβουλίο μας. Όταν βγαίνει και λέει ο Επίτροπος ότι συμφωνώ με την κριτική αυτή, θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι καλή η πρόταση και θα ήθελα μαζί από κοινού με εσάς, ως Επιτροπή, ως Κοινοβούλιο, να αναδιαμορφώσουμε την ε, πρόταση αυτή προκειμένου να ξεχωρίσουμε τα θέματα διαφήμισης και ασθενών. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι πάρα πολύ ουσιώδες, έχουμε τεράστια ευκαιρία μπροστά μας την οποία δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Αυτό θα σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια μεγάλη, να πάρουμε στα σοβαρά τη διαδικασία αυτή, αλλά να προσπαθήσουμε επίσης να βρούμε και μια ευρεία συνένεση και γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλό το είπε ο Κρίστοφερ Φιέλνερ ε, ότι δεν υπάρχουν ε, ιερές, αν θέλετε, τροπολογίες, όλα είναι υπό διαπραγμάτευση. Αν καταφέρουμε να βρούμε μια ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος Ντάλι, γιατί έρχεται πάντα στην πρώτη ανάγνωση, Το ξέρετε ότι σηκώνεται ο Επίτροπος και λέει συνήθως ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, βελτιώνουν την καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιες άλλες δυστυχώς θα πρέπει να τις απορρίψουμε. Αυτή είναι δυστυχώς η διαδικασία που ήθιστε. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι στην περίπτωση αυτή ο Επίτροπος θα τονίσει ότι ακριβώς οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου είναι αυτές οι οποίες βελτιώνουν και κάνουν καλό το κείμενο. Φυσικά πολλά θα πρέπει ακόμα να συζητήσουμε γιατί εξαρτώμαστε και από το νομικό συμβούλιο, αλλά από πολιτικής απόψης πραγματικά θα ήταν ανόητο να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία για να συγκαθορίσουμε, αν θέλετε, ένα τόσο σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω τώρα για την έκθεση συγκεκριμένα τον Κρίστοφερ Φιέλνερ. Συμπεριλέλαβε πολλά στοιχεία τα οποία είναι ουσιώδη και που βελτιώνουν σαφέστατα την κακή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο βάζουμε τον ασθενή και δεν ε, είναι το θέμα το ότι επιτρέπεται να κάνει η βιομηχανία. Μιλάμε για την διάθεση τη διθεσιμότητα πληροφοριών, αν θέλει ο ασθενής ε, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν του παρέχονται χωρίς να το ζητήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί μια φαρμακοβιομηχανία αφιερώνει μία ολόκληρη σελίδα σε διαφημίσεις σε μία εφημερίδα. Γιατί να κλείνει έτσι μια ολόκληρη σελίδα σε μια εφημερίδα ή σε διάφορα άλλα σε, ε, έντυπα αν δεν έχει συμφέρον, αν δεν πουλάει τελικά. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό το διαγράφει ο εισηγητής, συμφωνήσω και ο κύριος Χατζημαρκάκης, αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα θετικό. Οι πιστοποιημένες ε, πληροφορίε, νομίζω ότι αυτό είναι διαφυσβέτητο. Θα πρέπει να διατίθενται, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο. Γιατί πολλές φορές ένα ασθενή θέλει πληροφορίες, θέλει αυτό το σημείωμα που εσωκλείεται στα φάρμακα σε μια άλλη γλώσσα από την ε, επίσημη γλώσσα της ε, χώρας. Για παράδειγμα, στον Νοτιό Τυρόλο, όταν, για παράδειγμα, τίθεται θέμα μειονοτικής ε, γλώσσας. Γιατί να μην διατίθενται αυτέ οι πληροφορίε χωρί κανένα περιορισμό. Πρόκειται για εγκεκριμένε πληροφορίε. και φυσικά θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το ισοκλειόμενο σημείωμα να είναι πιο ευανάγνωστες και κατανοητές ε, οι πληροφορίες. Περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία στην έκθεση αυτή και περιλαμβάνονται και στοιχεία στην έκθεση της κυρίας Μακέβαν για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Και εκεί αναφέρονται οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο σου αυτό σημείωμα και θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και στην έκθεση της Λίντα Μακέβανς. Ε, ένα δύσκολο θέμα υπάρχει και στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γιατί δεν είναι απλό. Τι θα κάνουμε με το διαδίκτυο. Εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη λύση θα ήταν και στο ίντερνετ να δημοσιεύονται οι πιστοποιημένες πληροφορίες. Υπάρχουν όμως κάποιες ε, ε, χώρες που έχουν συνταγματικές αμφιβολίες και στη δική μου χώρα συζητιέται το θέμα αυτό, όχι τόσο έντονα όμως όσο στη Σουηδία. Και εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι νομικός, αλλά από ό,τι άκουσα και από την έκθεση Μικολάζικ, ε, μπορεί και να ρωτήσει κανείς τρεις ε, νομικούς και να πάρει τρεις ε, διαφορετικές απόψεις, μην σας πω και τέσσερις. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι τα, οι νομικοί έχουν διαφορετική αντίληψη, αλλά δεν θεωρώ ότι νομικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει έλεγχος των πληροφοριών που διατίθενται μαζί με ένα φάρμακο στο διαδίκτυο. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχει απαγόρευση σε κάποιες χώρες. Για να είναι λοιπόν λιγότερο αυτή, αυτή η απαγόρευση, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για λογοκρισία όταν ελέγχουμε το ισοκλειόμενο αυτό μήνυμα στα φάρμακα. Απλά ελέγχουμε κατά πόσο δεν, προκαλούνται, δεν προκαλείται κάποια ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι πιστοποιημένες πληροφορίες δεν είναι επικίνδυνες. Και αν αυτό ελέγχεται διαρκώς, εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να προκληθεί κάποια χειραγώγηση. Στην Σουηδία μπορεί να λειτουργεί το σύστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το σύστημα ή θα λειτουργούσε και στις άλλες 26 χώρες ε, μέλη. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό θα θέλαμε να το κοιτάξουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Κατά τα άλλα να πω ότι η έκθεση, το σχέδιο αποτελεί καλή βάση για την περαιτέρω εργασία μας και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συνεργασία για να καταλήξουμε σε μια αυρία συμφωνία. Ε... Ευχαριστούμε τον Πέτερ. Ο κύριος Ταραμπέκερ θέλει να παρέμβει εκ νέου. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να προσθέσω στην προηγούμενη μου παρέμβαση ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κ. Σουχένιε στην έκθεσή του παραδέχεται τα προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι υπάρχουν κοινά σημεία στο, στην εκκίνηση και νομίζω ότι με την επανεξέταση αυτή από τον νέο επιτρόπο, τον κύριο Νταλή, δημιουργείται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακριβώς κάποιες σκέψεις και ιδέες που υπάρχουν στο σχέδιο οδηγίας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και γι' αυτό η Κομισιόν ε, βλέπει με πολύ θετικό πνεύμα την περιττέρω διαδικασία και δεν θέλω να ευχαριστώ εδώ επί συγκεκριμένο σημείο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βάις Γκέρμπερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα κάτι να πω για το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Θα ήθελα καταρχήν να εγκομιάσω τον εισηγητή, γιατί πιστεύω ότι ε, έχει πάρα πολύ θετικά σημεία. Νομίζω ότι η έκθεση θα είναι πάρα πολύ θετική, πάρα πολύ ισορροπημένη. Ακούσαμε διαμακρών αυτό το θέμα της ενημέρωσης των ε, ασθενών και χαίρομαι που η ριζική αντίσταση που υπήρχε αρχικά κατά τις πρόσθεσης Κομισιόν τώρα τροποποιείται και οδηγείται σε μια επικοδομητική συζήτηση. Γιατί λέμε ότι εντάξει, συζήτηση, την πρόταση Κομισιόν όσο έχει δεν τη θέλουμε, αλλά θέλουμε συγκεκριμένα βελτίωση τη ενημέρωση των ασθενών και θέλουμε να πετύχουμε τον ενήλικο όριμο ασθενή όπω θέλουμε τον ενήλικο και όριμο καταναλωτή. Και γι' αυτό είμαι θετικά διακείμενη και πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Αναφέρθηκαν σημαντικά σημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξαιρέσουμε τα ε, έντυπα μέσα ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να ελέγχεται εκ των προτέρων η πληροφόρηση που δίνεται, αλλά τελικά εάν ε, λάβουν υπόψη σοβαρά το σημείο αυτό και κάποια άλλα σημεία ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι ο ασθενή και όχι η βιομηχανία, ότι δεν θα έχουμε διαφήμιση αλλά ενημέρωση για τον ασθενή. Όλα αυτά θα καταστήσουν την πρόταση προ όφελο του ε, γιατί Γιατί ομολογώ, όταν πηγαίνω εγώ στο γιατρό και θέλω κάποιες πληροφορίες, ο γιατρός δεν είχε αρκετό χρόνο και εγώ θέλω να ενημερωθώ ίσως εκ των υστέρων, αλλά καμιά φορά και από πριν. Αλλά τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κάποιε πληροφορίε στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι καλή ποιότητα, δεν έχουν ελεγχθεί. Και όταν ακούω ότι το Συμβούλιο λέει ότι δεν χρειαζόμαστε ε, νομοθετικές πράξεις γιατί υπάρχουν ήδη πολλέ πληροφορίε στο διαδίκτυο, εγώ λέω όχι. Όχι, γιατί μια θέση πληροφορίες δεν είναι καθόλου καλέ. Και οι γιατροί μου λένε ότι χρειάζονται 10 λεπτά για να αντιστρέψουν τις κακές πληροφορίες που είχε ο ασθενή σε καλές. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θέλουμε ανοιχτά προσβάσιμες καλές και ελεγμένες πληροφορίες. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικά σημεία. Καταρχήν η πληροφορία στο συνοδευτικό φυλάδιο των φαρμάκων που θα μπορέσει να προσφέρεται και από τη βιομηχανία στην ιστοσελίδα ε, της. Και από την άλλη χρειαζόμαστε μια γενική ιστοσελίδα που θα δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες για διάφορα φάρμακα ή βασιζόμενη στις ασθένειες να δίνει τις πληροφορίες αυτές στους ασθενείς. Δηλαδή να μπορεί να ενημερωθεί ο ασθενή όχι μέσω τη ιστοσελίδα τη εταιρεία μονάχα, αλλά ε, να, εξετάζει βάση τη ασθένεια που έχει. Α πούμε, έχω ψηλή πίεση. Κοιτάει στην ιστοσελίδα και κοιτάει τι γίνεται. Γιατί εκεί θα λέγονται όχι μόνο τα φάρμακα που χρειάζονται, αλλά και η υγιής ε, ε, διατροφή, σπορ κλπ. Κάτι παρόμοιο υπάρχει ήδη στο, στην Σουηδία, μόνο που ξεκινάνε μάλλον από τις ασθένειες, αλλά από τα φάρμακα. Και θα έλεγα ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλουμε ένα μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι θα θέλαμε να υπάρχουν στα κράτη-μέλη τέτοιου είδους στοιχεία. Όχι σαν ευρωπαϊκή λύση, αλλά στα κράτη-μέλη ίσως, αποκεντρωμένα. Θα ήταν καλό να είχαμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων και έχουμε τη σωστή συζήτηση για το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Κανένας άλλος δεν ζητάει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τους στόχους. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει καλή μορφή. Προσπαθούμε να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο για να μπορέσουμε να εργαστούμε επικοδομητικά, να συνεργαστούμε με την Επιτροπή. Ε, δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι παρευρισκόμενοι είναι δύσκολο λοιπόν να αποφασίσουμε εμείς μεταξύ μας. Προτείνω λοιπόν να το αφήσουμε για αύριο το πρωί για τους συντονιστές οι οποίοι αν το επιθυμούν θα, θέσουν ξανά, θα μας θέσουν ξανά το ερώτημα στις 10 δηλαδή μετά τη συνάντησή τους για να εργαστούμε όπως πρότειναν μερικοί, δηλαδή οι σκιώδεις, να συναντηθούν με τον εισηγητή για να έχουμε μια πιο εύρωστη πρόταση ή ενδεχομένως να το αναπέμψουμε για αργότερα. Οι συντονιστές θα το αποφασίσουν και μετά θα δούμε κατά πόσο θα, θα συμφωνήσετε όλοι, θα συμφωνήσουμε όλοι μάλλον. Ε, ευχαριστώ λέει ο εισηγητής. Εκπλήσουμε κάπως. Uh, and, and I strongly dislike, but this, I strongly dislike when interesting, important and... Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν αντιγνωμίες δεν πρέπει να αποτελέσουν μία γραφειοκρατική διαδικασία και μόνο. Ακούσα διαφορές μεταξύ σοσιαλιστών και πρασίνων σε πολλά επίπεδα. Αλλά η άποψη των σοσιαλιστών ήταν κάτι το νέο για μας. Ε, λυπάμαι που θα απορρίψετε αυτό θα περίμενα να το ακούσω από την Ισπανική Προεδρία ή από το Συμβούλιο, αλλά όχι από τους σοσιαλιστές. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε προετοιμάσει μια τέτοια, προετοιμάζουμε μια τέτοια πρόταση κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια. οι σοσιαλιστές συνάδελφοι είπαν ότι ο επαγγελματικός κλάδος θα πρέπει να δώσει μία λύση. Αυτό το κατέγραψα και το αναφέρω και στην έκθεση. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη από πλευράς ασθενών. και τρώγοντας έρχεται η όρεξη, για να το πω και έτσι. Πολλοί ασθενείς ψάχνουν στο διαδίκτυο κάθε μέρα και λαμβάνουν ε, αβέβαιες, ανασφαλείς πληροφορίες. Το ξέρουμε σαν γεγονός. Γι' αυτό θα πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό ε, το ζητάμε κατεπηγόντως και από τις ενώσεις ασθενών έμαθα ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ασθενής. Οι ασθενείς είναι όλοι διαφορετικοί. Εγώ πάσχω από χρόνιο άσθμα και νομίζω ότι μπορώ να διαχειριστώ ορισμένες πληροφορίες για την ασθένεια με την οποία ζω εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν όμως σπάνιες ασθένειες όπου οι πληροφορίες δεν είναι τόσο πολλές. Στην ιατρική υπηρεσία, όταν, ε, βρέθηκα, όταν χρειάστηκε να πάω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ε, έδειξα το μηχάνημα που χρησιμοποιώ, είδα ότι ο γιατρός μπήκε στο Google για να δει τι είναι αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιώ, δεν το ήξερε. Ελπίζω να βρει και τη σωστή πηγή, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάμε και γιατί ξεκινήσαμε. Το ξέρω ότι δεν είναι μια ολοκληρωμένη λύση. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας και να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα σωστά ζητήματα, δηλαδή να το βλέπουμε το κάθε θέμα σημείο προς σημείο. Χαίρομαι για την άποψη της Επιτροπής, διότι ακριβώς αυτό είπα και στον κύριο Ντάλι, στον Επίτροπο. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. είπε ότι θέλει να ακούσει την άποψη των ασθενών, να έχουμε την οπτική γωνία των ασθενών. Αυτό προσπάθησα να κάνω, να τα δω όλα υπό το πρίσμα των ασθενών. Αυτή είναι μια εξαιρετική ε, ευκαιρία που έχουμε να επηρεάσουμε την Επιτροπή. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε την ε, πρόταση, μα ακριβώς αυτό κάνουμε. Η κυρία Χάση είπε ότι ίσως υπάρχουν άλλοι τρόποι να διαδώσουμε την άποψή μας, αλλά ο παραδοσιακός τρόπος είναι να συζητήσουμε, να τροποποιήσουμε, να αναθεωρήσουμε, να φτάσουμε σε ένα συμβάσμα. Μη μου πείτε ότι χρειάζεται μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Την ίδια οδό θα ακολουθήσουμε και τότε. Και δεν έχω χρόνο μπροστά μου. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να περάσει αυτό το θέμα. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο το πρωί, να το συζητήσουν οι συντονιστές. Μη μου πείτε όμως ότι πρέπει να παρετηθούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας ως προς αυτά που είπατε. Όλοι συμφωνούμε από όλες τις πλευρές, από όλο το πολιτικό φάσμα, ότι θα πρέπει να έχει ο ασθενής όλα τα μέσα στη διάθεσή του για να μπορεί να αποφασίσει. Γίνεται μία συζήτηση. Εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ απόψη, γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Οι παρευρισκόμενοι δεν θέλουμε να το αναπέμψουμε στις ε, καλένδες. Απλώς, αύριο το πρωί οι συντονιστές θα δουν τι πρέπει να γίνει, δεν θα χάσουμε χρόνο και θα μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε το αργότερο, το αργότερο αύριο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πώς θα το διευθέτησουμε, αυτό σας προτείνω. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση, η λιγότερο κακή εν πάση περιπτώσει, γιατί ο χρόνος τρέχει. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ λέει και ο εισηγητής. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα, που αφορά την έκθεση επί της ανακοίνωσης επιτροπής για την κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και δίνω το λόγο στον Ζουάου Φερέιρα που είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. τα πρόσφατα γεγονότα, οι καταστροφές στη Μαδέιρα, στη Γαλλία δείχνουν ότι το θέμα είναι επίκαιρο και σημασία έχει η πρόληψη. Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την σημασία αυτού του θέματος. Και επίσης επιβεβαιώνει κάτι το οποίο γνωρίζαμε ήδη κατά τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του ε, Ταμείου ε, Αλληλεγγύης η Επιτροπή έλαβε 62 αιτήσει από 22 διαφορετικές χώρες για οικονομική αρρωγή. Όταν ε, τουλάχιστον μιλάμε για καταστροφές μεγάλων φυσικών διαστάσεων. Χρειάστηκε λοιπόν κινητοποίηση του Ταμείου αν και δεν μπορέσαμε να δράσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι οι ζημιές δεν μπορούν να ποσοστοποιηθούν και, εν πάση περιπτώσει, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αντίτιμο. Αυτό το ξέρουμε. Σε αυτά τα πλαίσια η πρόληψη θα πρέπει να έχει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία μέσα στα πλαίσια του κύκλου διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουν καταρχήν τους πολίτες τους και να προλαμβάνουν τις φυσικές καταστροφές στο μέτρο του δυνατού. Αλλά θα πρέπει να επαυξηθεί και η συνεργασία και καλύτερος συντονισμός μεταξύ κρατών μελών και Ταμείου Αλληλεγγύης. Άρα η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβάλλει ορισμένες νέες προτάσεις και αυτό που έχει σημασία είναι να κινηθούμε πέρα πέραν της ανακοίνωσης. Υπάρχει ένα σύνολο δράσεων που θα προβάλλει η Επιτροπή και που προβάλλει μέσω της ανακοίνωσης και τόσους μήνες μετά αυτά τα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν. Υπέβαλα ερωτήσεις προς την Κομισιόν και γραπτός και προφορικά και χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα και η Γενική Διεύθυνση Προστασίας των Πολιτών Η Επιτροπή ε, όρισε τρεις κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες όμως δεν δόθηκε συνέχεια. Η ιεράρχηση πληροφοριών για τις ε, φυσικές καταστροφές, διενέργεια μελέτης για τις ε, πρακτικές χαρτογράφησης των κινδύνων στα κράτη-μέλη και με βάση αυτή την έρευνα κατευθυντήριες γραμμές χαρτογράφησης των κινδύνων και τέλος, ένας απογραφικός κατάλογος των ε, κοινοτικών μέσων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εργασία πρόληψης. Έχω λάβει απάντηση μόνο στο τελευταίο ερώτημα, γιατί στο μέλλον έμαθα ότι θα υπάρξει αυτός ο απογραφικός κατάλογος, θα διενεργηθεί αυτή η μελέτη. Αναμένουμε τα στοιχεία κατά τα τέλη Ιουλίου. Αν έχουμε αυτά τα στοιχεία, αυτό θα μας ε, βοηθούσε ιδιαίτερα για να προετοιμάσω καλύτερα και την έρευνα, αλλά η ενίσχυση αλληλεγγύης μεταξύ κρατών ε, μελών επιβάλλεται και επιβάλλει ε, μια σωρία μέτρων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και πρόληψης όπως προτείνει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στην έκθεση πάμε και λίγο παραπέρα ως προς τη συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο, όπου θα συμμετέχουν και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές. Αυτό προέβαλε και η Γενική Διεύθυνση Ρέτζι, έτσι ώστε να γνωρίζουμε λεπτομεριακά τις τοπικές συνθήκες. Αυτό το δίκτυο θα αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και ανείχνευσης αιτιών που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Θα πρέπει να, να συμμετάσχουν και κοινωνικές οργανώσεις Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το μέγεθος των ε, καταστροφών. Δεν μιλάμε όμως μόνο για φυσικά φαινόμενα. Πολλές φορές ε, οι καταστροφές ε, υπόκεινται σε κακοδιαχείριση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ε, οφείλεται σε ε, χωροταξικά σχέδια, σε μη σωστή διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και ανακύπτουν πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το στοιχείο ευαλωτότητας, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές που πλήττονται πολύ συχνά. Θα πρέπει λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και το χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο θα χρησιμοποιήσει τα ήδη προϋπάρχοντα μέτρα, ιδιαίτερα ως προς την περιφερειακή πολιτική που και πολιτική περιβαλλοντικής και περιφερειακής ανάπτυξης θα πρέπει να προβάλλουμε μέτρα καθαρά πρόληψης που να τύχουν προτιμησιακής χρηματοδότησης διότι οι φυσικές καταστροφές έχουν πλήξει πολλά κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε λοιπόν μία σειρά κοινών δράσεων για αυτή την ε, χρηματοδοτική πλαισίωση. Δεν ε, εξαντλώ το όλο ζήτημα, αλλά σας προβάλλω έναν ενδεικτικό κατάλογο μέτρων, αναγκαίων μέτρων, μετά από τις ε, πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Μιλώ για διόρθωση καταστάσεων που οδηγούν σε κίνδυνο ή σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, να προστατεύσουμε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν είναι ευάλωτες, να ελέγξουμε τα δίκτυα ασφάλειας των έργων υποδομής, και να δούμε κατά πόσο γίνεται σωστή χρήση της γης. Επίσης θα πρέπει να ενσωματώσουμε το σκέλος της πρόληψης στον προγραμματισμό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναδιατυπωθούν προγράμματα εκεί όπου χρειάζεται στα κράτη-μέλη. Επίσης, αναγνωρίζουμε και τις ανάγκες των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών ή των αρεοκατοικημένων περιφερειών. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε έναν ιερχικό κατάλογο, έναν απογραφικό κατάλογο των αναγκών, ιεραρχώντες της και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ε, συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι γνωρίζουν πολύ καλύτερα την ε, τοπική πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, ένα σωστός διάβλος χρηματοδότησης μέσα στα πλαίσια αυτής της δικτύωσης και να μην κινούμαστε μόνο με βάση κοινά, κέντρα, κοινά ερευνητικά κέντρα. Με βάση τα κοινά ερευνητικά κέντρα, τα οποία πολλές φορές έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα. θα πρέπει να προβάλλουμε μέτρα προσαρμογής ως προς τον αστικό ιστό και τον, ε, τον αστικό ιστό και τον ιστό της υπαίθρου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα ακραία κλιματικά φαινόμενα και να προσπαθήσουμε να μικρύνουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών, ιδιαίτερα ως προς τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες και να ορίσουμε περιφέρειες υψηλού κινδύνου, να τις αναγνωρίσουμε, να τις ε, ταυτίσουμε μέσα στα πλαίσια της ε, πρόληψης. και οι φυσικές καταστροφές δυστυχώς πλήττουν κατά κανόνα αυτούς που διαθέτουν ε, λιγότερους πόρους. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ορισμένα είδη φυσικών καταστροφών που ανακύπτουν συνέχεια. θα πρέπει να συσταθεί ένα παρατηρητήριο και μία πρωτοβουλία για την προστασία των ε, δασών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης Προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να συμπεριλάβω όλα τα στοιχεία που ε, θα θέλατε, καθώς και τα στοιχεία που έλαβα από την Ρέτζη και την Επιτροπή ε, Γεωργίας. Και έλαβα υπόψη και άλλα στοιχεία στα οποία δεν είχε δοθεί συνέχεια μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. για ένα σημείο το οποίο μας απασχολεί όλους. Θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. ξεκινώντας από την κυρία Εστρέλα. Αυτό είναι ένα θέμα ζωτικής ε, σημασίας και νομίζω ότι η παρέμβαση της Επιτροπής ε, έγινε την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία αυτή. Είναι ένα θέμα που ανακύπτει συνέχεια στις συζητήσεις μας. Ξέρετε τι συνέβη πολύ πρόσφατα στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Η φυσική καταστροφή στη Μαδέρα, στην Γαλλία, στην Ισπανία και σε τρίτες χώρες όπως στην Αϊτή, στη Χιλή. Αυτό που έχει σημασία είναι να ασχολούμαστε έγκαιρα με αυτά τα ζητήματα, προσπαθώντας να εξεύρουμε λύσεις και να ορίσουμε επαρκείς ε, πολιτικές για να προλάβουμε τις ε, φυσικές καταστροφές εκεί που, όπου μπορούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όποτε ανακύπτουν, να έχουμε τουλάχιστον τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης. Να ε, μην υπάρχει να μην υπάρχουν μεγάλες ζημιές και να μην χάνονται και ανθρώπινες ζωές βεβαίως κυρίως. Οι φυσικές καταστροφές σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και γι' αυτό πιστεύουμε ε, δυστυχώς ότι θα ανακύπτουν όλο ένα και περισσότερο. Στο μέτρο της πρόληψης Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Σας θυμίζω ότι το 2006 ήμουν η συγγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, επί του θέματος αυτού, όπου ε, τόνιζα την ανάγκη λήψης μέτρων ιδιαίτερα για την πρόληψη και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της έρευνας και άλλα μέτρα τα οποία, στα οποία δώσε συνέχεια τώρα ο εισηγητής. Εκεί όπου δεν δόθηκε δηλαδή ικανοποιητική απάντηση σε σχέση με τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε. Τα θέματα αυτά είχαν ε, εκφραστεί ήδη από το 2006 ιδιαίτερα για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ξηρασία και την απερίμωση. Πρόσφατα, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία αυτού, του παρατηρητηρίου Τα μέτρα όμως αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. γιατί θα ζούμε ε, ολοένα και μεγαλύτερης περίοδους ξηρασίας με πυρκαγιές και με μεγάλες πλημμύρες. είναι ένα θέμα που πλήττει ιδιαίτερα την ε, κεντρική και νότια Ευρώπη. Δυστυχώς το Σεπτέμβριο όταν ε, επανήλθαμε στις ε, εργασίες μας μιλήσαμε για τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, μιλήσαμε για καλές προθέσεις, αλλά δεν έγινε τίποτα άλλο. θα υποβάλω κι εγώ μία έκθεση, διότι χρειάζεται μία οδηγία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Υπάρχει μία οδηγία για τις πλημμύρες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε συντάξει ακόμα μία οδηγία για, την αντιμετώπιση των ε, πυρκαγιών. Μιλάμε για εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ε, πρόληψη και για την έγκριση καλών πρακτικών Και δεν μπορώ να ξεχάσω την ε, ανάγκη σύνταξη μιας τέτοιας οδηγίας. Δυστυχώς έχει ε, μπλοκάρει η νέα πρόταση ε, απεμπλοκής του Ταμείου Αλληλεγγύης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό θα πρέπει να απεμπλακεί αυτή η κατάσταση ως προς το Ταμείο Αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις, έκρηθμες καταστάσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, πυρκαγιών καλύτερα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον φυσικό μας πλούτο, ιδιαίτερα τα δάση. Και θα πρέπει να μπορούμε να δούμε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τη, τις εκτάσεις αυτές, τις γέες αυτές, οι οποίες έχουν απεριμωθεί. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ευθύνη Το θέμα αυτό επήγει, έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα και εδώ θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να χαρτογραφήσουν τους κινδύνους σε σχέση και με τις πλημμύρες αλλά και με τις πυρκαγιές έτσι ώστε να τις προλαμβάνουμε όπου μπορούμε. Je Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόταση που είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Το λόγο έχει ο κύριος Ούγκιας. <clears throat> Oh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερέιρα για την εξαιρετική αυτή εργασία. Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο από το να καταγράφουμε καταστάσεις μετά από τις καταστροφές στη Μαδέρα, στα Κανάρια νησιά, στην Ανδαλουσία. Είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος. Και ε, όπως είπε και ο συνάδελφος Αλφονσίν, ε, χτες επλήγει η Σικελία, η Ιταλία, αύριο μπορεί να πληγεί μια οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιφέρεια. Θα πρέπει να αναλαμβάνουμε λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δίνουμε συνέχεια στα θέματα αυτά. Θα πρέπει, όπως ε, αναγράφεται στο σημείο 5, να σταθούμε ιδιαίτερα στους πόρους και να έχουμε ένα επαρκές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Γιατί αν δεν γίνουν επενδύσεις, δυστυχώς θα πρέπει στη συνέχεια να μας απασχολήσει υπό μορφή αποζημιώσεων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό ακριβώς να μας απασχολήσει. Θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής όλες οι κατευθυντήριες γραμμές, οι κατευθυντήριες γραμμές που αναγράφονται εδώ, θα πρέπει να περάσουν από ένα αριθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο προγραμματισμού. Γιατί εδώ εμπλέκονται και δημόσιοι φορείς. Θα ήθελα να σας πω ότι θα υποβάλω μία τροπολογία επ' αυτού, δηλαδή σε κάθε γενικό προγραμματισμό των ε, περιφερειακών διαμερισμάτων να υπάρχει ένα κεφάλαιο που να αναφέρεται σε δαπάνες πρόληψης. Δηλαδή σε κάθε προϋπολογισμό περιφέρειας, περιφερειών, σε κοινοτικό ή δημοτικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δαπάνες πρόληψης, έτσι ώστε κάθε κοινότητα να ξέρει τι δαπάνες προβλέπονται, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές στο μέτρο του δυνατού. Βεβαίως, ε, ως προς τα τσουνάμι, τους σεισμούς ε, δεν μπορούν να προληφθούν. Ο Νικολό Μακιαβέλη είχε αναφερθεί σε αυτό το θέμα και είχε πει ότι τα ποτάμια πλημμυρίζουν πάντα, αλλά όταν ε, προβάλλουμε συγκεκριμένα έργα και φράγματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα αυτή την υπερχείληση. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο αντιμετώπισης της ξηρασίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 16 Ιουνίου θα γίνει μια συζήτηση για το, το πρόγραμμα GMES και εδώ υπάρχουν ε, διάφορα μέσα που προβάλλονται ως προς, αυτή την, ε, ως προς αυτές τις δραστηριότητες για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το μέσον. Εδώ θα πρέπει να ενσωματωθούν, να ενταχθούν αυτά τα μέσα. Θα πρέπει δηλαδή να ενταχθούν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα στο ΟΓΜΕΣ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ζαν Μάρη. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και πολύ καλό και ισορροπημένο το κείμενο, το σχέδιο έκθεσης του κ. Φερέιρα. Έχει καλύψει τα πιο σημαντικά από τα ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, το χωροταξικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, τη χαρτογράφηση των κινδύνων και τα ζητήματα χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει πιο δυνατό μέσα στο κείμενο είναι το ζήτημα της κοινή μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση των κινδύνων και των καταστροφών. Μπορούμε να αναζητήσουμε πιο δεσμευτικές λύσεις από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ένα ελάχιστο επίπεδο χαρτογράφησης που θα πρέπει να αναλάβουν έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο εναρμονισμένο και πιο αποτελεσματικό σύστημα. Βεβαίως και συμφωνούμε στην ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη των καταστροφών για την περίοδο μετά το 2013. Θα θέλαμε όμως πιο αποτελεσματική αξιολόγηση των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων με ταυτόχρονη επιτήρηση και έλεγχο από τις ευρωπαϊκές αρχές για την ορθή αξιοποίηση αυτών των ε, κονδυλίων. Θα μπορούσαμε μάλιστα να προσθέσουμε και δικλείδες ασφαλείας, το έχει ξανακάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε καταγεγραμμένη περίπτωση μίσος της αξιοποίησης των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη, να διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να τις επιστραφούν αυτά τα κονδύλια. Θυμίζω ότι μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε μια τέτοια πρόταση που αφορούσε την ε, περίπτωση τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δουν για αλληλεγγύη, για αποκατάσταση των καμένων περιοχών στον ε, Ευρωπαϊκό Νότο αν αυτές οι ε, εκτάσεις οικοπεδοποιηθούν ή τουριστικοποιηθούν να επιστρεφούν τα χρήματα. Μέσα υπάρχουν βεβαίως και κάποιες δυνατότητες για παραπέρα δυνατού, όπως ε, εκεί που μιλά για τα αντιμετώπιση των γενσιουργών παραγόντων των κινδύνων ε, έχει κάπου τη φράση για χωροταξική αναδιάταξη των δασών. Αυτό αφήνει κάποια περιθώρια ε, να μην χρησιμοποιηθεί με αηφορικό τρόπο αυτή η αναδιάταξη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνει έμφαση στην αναδάσωση για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, όταν μιλά για να δοθεί έμφαση στα φράγματα, θα πρέπει να προσδιοριστούν. Να μιλήσει, προτείνουμε, για μικρά φράγματα ανάσχεσης της ροής των ε, νερών, ούτε ώστε να προλαβαίνουν να απορροφώνται στα πιο ορεινά σημεία και να μην ε, αυξάνεται η ποσότητα ε, που τελικά καταλήγει να δημιουργεί προβλήματα. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, αν και η συγκεκριμένη έκθεση μιλά για την πρόληψη, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια αναφορά στην έκθεση Μπαρνιέ σχετικά με την ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας και τη διασύνδεση της πρόληψης με την αντιμετώπιση των ε, φυσικών καταστροφών. Είναι πάντως ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο και εμείς θα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιανακουδάκη. Thank um, θα ήθελα να διαβάσω ένα κείμενο εξ των σκιωδών των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Φερέιρα για την έκθεση. Όπως προτείνει και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε μία ε, αύξηση φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία ώστε τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να συνδράμουν για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και να υποστηρίζουν τους πολίτες εκεί που δεν προλαμβάνονται. Θα πρέπει να προσδοθεί μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Επίσης, χρειάζεται δράση σε κοινοτικό επίπεδο μαζί με το εθνικό και μία ε, κοινή προσέγγιση εκεί όπου χρειάζεται. Κατά την άποψή μου το σχέδιο έκθεσης ε, κινείται πέρα από τη συμπλήρωση των εθνικών δράσεων. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιο κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να οικοδομηθεί με βάση μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τα προϋπάρχοντα κοινοτικά μέσα για την πρόληψη δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο όπως προτείνει ο εισηγητής. Η πρόληψη αφορά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και η δράση σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές δράσεις. Ευχαριστώ. Je vous Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καρσία. Sí, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί στην Επιτροπή Γεωργίας συζητούσαμε μία σημαντική εκθέση και δεν μπορούσα να βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερέιρα για τις ιδέες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή του και γιατί τονίζει την ανάγκη βελτίωση συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, σε κοινοτικό και εθνικό, καθώς και περιφερειακό. Οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα και θα πρέπει να τύχουν συνολικής αντιμετώπισης. Μπορούμε να έχουμε μία πλημμύρα στη Γερμανία ή ε, μία ε, πυρκαγιά στην Ελλάδα ή στην Ιβηρική Χερσόνησο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την κατάλληλη πρόληψη χωρίς διακρίσεις ως προς τη συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους τομείς για να έχουμε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία ήδη προϋπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο. Ως προς την πρόληψη φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Συμφωνώ με τον εισηγητή και θα υποβάλω μία σειρά τροπολογιών. Θα πρέπει να δράσουμε εξ άντε και εξ post και να υπάρξει μία οδηγία κατά της ξηρασίας όπως ισχύει κατά των πλημμυρών, διότι οι παρατηνόμενες ξηρασίες γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες και αυτό το γνωρίσαμε στην Ισπανία, σε ένα μεγάλο μας ε, φυσικό πάρκο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, να την εξατομικεύουμε. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε και το ρόλο του αγρότη, του θεματοφύλακα της υπαίθρου και η γεωργική δραστηριότητα να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και να μην απεριμόνονται οι περιοχές, διότι αυτό θα σήμαινε κοινωνική και περιβαλλοντική καταστροφή αν εγκαταλείψουμε την Υπέθρο. Στον τομέα των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εισαγάγει μία πραγματική δασονομική πολιτική για την διατήρηση των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των δασών που είναι πραγματικοί πνεύμονες. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση και την ξυλία μας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να διαθέσουμε ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο προσαρμογής των διαφόρων τομέων για να προλαμβάνουμε φυσικές καταστροφές στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσω να συνδράμω και εγώ στην ενδιαφέρουσα έκθεση του κυρίου Φερέιρα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα το λόγο το... στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Le, le rapporteur pour son avis, ainsi que le Parlement européen qui s'est exprimé euh, très régulièrement. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι έχει μιλήσει επί μακρόν στο θέμα της πρόληψης. Έχουμε τι προσέγγιση, θέλουμε να ανταποκριθούμε στις καταστροφές, αλλά μας ενδιαφέρει και το σκέλος της πρόληψης, να υπάρχει αλληλεγγύη δηλαδή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, βεβαίως να τονίσουμε και την αρχή της ευθύνης ως προς την πρόληψη. Από την έγκριση αυτής της ανακοίνωσης, η Επιτροπή έχει προβάλει ορισμένες ε, δράσεις που υπενθύμησε και ο εισηγητής ε, για να γνωρίζουμε τις καταστροφές, να τις χαρτογραφήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, η ανάλυση κινδύνων, όπως υποστήριξε και ο εισηγητής. Θα θέλαμε η πρόληψη να ενσωματωθεί καλύτερα στα χρηματοδοτικά μέσα που προϋπάρχουν. Γι' αυτό διενεργήσαμε μία μελέτη για τα διάφορα μέσα υποστήριξης και μας ενδιαφέρει η ύπαρξη καλύτερων συνδέσμων μεταξύ χρηματοδοτικού μέσου και πρόληψης φυσικών καταστροφών. Υπ' αυτή την έννοια θα ήταν αναγκαίο να ε, αναπτύξουμε μία μεθοδολογία για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, η Επιτροπή εργάζεται στο θέμα των δασών. Προετοιμάζουμε μία πράσινη βίβλο και αυτή η πράσινη βίβλος θα προβάλλει εναλλακτικέ για την πολιτική μας σε αυτό το θέμα ως προς το παρατηρητήριο κατά της ξηρασίας. Όπως είπαν και ορισμένα μέλη, εργαζόμαστε για τη συγκρότηση, για τη σύστασή του. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δώσουμε συνέχεια έτσι ώστε να γίνεται σωστή ε, ανείχνευση και ανταλλαγή δεδομένων. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Και εμείς ευχαριστούμε την Κομισιόν. Ξαναδίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Φερέρα, ευχαριστώντας τον για την ποιότητα αυτής της έκθεσης, όπως ε, ανέφεραν και όλοι οι ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, θέματα, αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε να γίνουν ε, και άλλες τροποποιήσεις. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και είμαι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μου αποστείλετε και γραπτός παρατηρήσεις και να συνεργαστούμε με τους σκιώδεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα θέμα που είναι ένα σημείο εκκίνησης. Μπορούμε να αποφύγουμε ορισμένες φυσικές καταστροφές, αλλά όχι τα ε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο δεν οδηγεί πάντα σε καταστροφή γιατί οι φυσικές καταστροφές πάντα θα υπάρχουν, υπήρχαν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. αλλά θα πρέπει να τις προλαμβάνουμε στο μέτρο του δυνατού. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω όλες τις παρεμβάσεις. Ως προς οδηγίες τώρα, Μιλήσατε για την οδηγία κατά της ξηρασίας και κατά των πυρκαγιών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο φυσικές καταστροφές. Ως προς την ξηρασία ίσως υπάρχουν ε, αντιγνωμίες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του θέματος Υπήρχαν και προγενέστερες συστάσεις, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λίγο καλύτερα τους ε, στόχους αυτού του παρατηρητηρίου. Ως προς την οδηγία κατά των ε, πυρκαγιών δεν προτείνεται μάλλον οδηγία, αλλά μία ειδική πρωτοβουλία της Επιτροπής για αυτό το θέμα των πυρκαγιών και της αναδάσωσης. υπάρχει ένα σοβαρό θέμα βιωσιμότητας των δασών. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη υλοτόμηση και όχι επαρκής αναδάσωση. Πρόκειται για μεγάλη μάστιγα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί λοιπόν μία εκτενής αναδάσωση, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες. προβάλλοντας την βιοπικιλότητα και την ε, αντιμετώπιση ασθενειών ε, ορισμένων ε, ειδών. Ως προς το χρηματοδοτικό πλαίσιο, είπε η συνάδελφος ε, ότι από τους ε, μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς ότι είπε ότι αντιτίθεται σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο. Εδώ δεν προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο. Αυτό που πρότεινα είναι να υπάρξει μία χρηματοδοτική πλαισίωση με βάση τα μέσα που προϋπάρχουν. Αυτή είναι και η άποψη των περισσότερων συναδέλφων και φαίνεται είναι, ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Δηλαδή πολιτική ε, συνοχής, μια πολιτική συνοχής μέσα σε μια χρηματοδοτική πλαισίωση. Η πρόληψη είναι πρωτογενής ε, υπόθεση των κρατών μελών. Αλλά αυτό που προτείνουμε είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Και θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έχουμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και προσπάθησα να ενσωματώσω και δικές τους υποδείξεις. Και θέλουμε να δούμε ποιες είναι και οι επιπτώσεις της ΚΑΠ, της ΚΑΠ στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Υπάρχει και εγκατέλειψη της υπαίθρου σε ορισμένες περιφέρειες. Άρα υπάρχει μεγάλη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα αυτών των ε, περιοχών. Θα πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια προσέγγιση αυτού του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη το σκέλος της πρόληψης. Αυτό το αναφέρω εκτενώς στην αιτιολογική έκθεση. Ο κύριος Τρεμόπουλος και ένας άλλος συνάδελφος ε, αναφέρθηκαν στα μέσα προγραμματισμού. Δηλαδή να έχουμε ένα κεφάλαιο, ειδικό κεφάλαιο για την ε, πρόληψη. Διότι είναι πρωτογενής ευθύνη των κρατών μελών. Αυτό ακριβώς λέμε όταν προτείνουμε την αναθεώρηση της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη την έγκυρη χρηματοδότηση. Επίσης θα πρέπει να γίνεται καλή χρήση των πόρων, βέλτιστη χρήση. θα πρέπει να πούμε ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί προβλέπουν επαληθεύσεις, ελέγχους. έτσι ώστε μέσω μηχανισμών επαλήθευση να δούμε κατά πόσο γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων. Αλλά στιγμή που δεν προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, δεν βλέπω γιατί ανησυχούν μερικοί. Bon, euh, euh, euh για τη διαθεσιμότητα πόρων και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ξέρετε ότι είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση. Μπορείτε να μου στείλετε τις παρατηρήσεις σας και γραπτός όποτε θέλετε, μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας, που θα μας αναγγείλει η Πρόεδρος. Είμαι στη διάθεσή σας. Merci, Σας ευχαριστώ διότι ε, πράγματι η προθεσμία είναι 22 Μαρτίου στις 12 στην ΕΜΒΗ θα ψηφίσουμε στις 4 ε, και 5 Μαΐου και μετά τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Χαίρετε.